Ε, προσβάλλει την εικόνα του Κοινοβουλίου. Επειδή εμείς προσπαθούμε εδώ να συνδυάσουμε η οικογένεια και δουλειά, ε, είναι λυπηρό και σχρόν ακούγονται τέτοιες φράσεις στο Κοινοβούλιο. Διότι εμείς αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε, την οικογένεια με τη δουλειά μας. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη πριν ψηφίσουμε. Θέλω να κάνω εδώ μερικές δηλώσεις. Ανακοινώσεις καλύτερα. Πρώτη, γραπτή δήλωση 007-2011 που παρουσίωσαν οι κύριοι Παπαστάμκος, Μπεναχμίας, Μίτσελ, Σούστα και Σύρκα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό και υπογράφηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου και αυτό είναι και ένα καλό νέο δηλαδή για τα τρέχοντα νέα που θολώνουν ε, την, αμαυρώνουν την εικόνα του αθλητισμού στην Ιταλία. Βάσει του άρθρου 123 του κανονισμού η ανακοίνωση θα δοθεί στους ε, παραλήπτες και θα δημοσιευτεί αντίστοιχα όπως επίσης <coughs> και τα ονόματα των βουλευτών που θα δημοσιευθούν στα πρακτικά. Γραπτή δήλωση 0010 του 2011 για να, για να Γκέριγκερ Όριμπερ, Γκρόστεκ, Γκρόστεκ και Βίνγκστρομ για τους εξαφανιστέντους, για τους αγνοούμενους στην Κύπρο που υπογράφηκε πλειοψηφικά από τα μέλη του Κοινοβουλίου και θα διαβιβαστεί βάσει του άρθρου 123 στους ε, παραλήπτες λοιπά Συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Ζήτησε σύντομα το λόγο. Η Μαρίνα Γιανακουδάκη ζητάει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. να είναι το όνομά μου. Τους τελευταίους τρεις μήνες στο γραφείο μου έστειλε ηλεκτρονικά μηνύματα, έκανε τηλεφωνήματα για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για αυτή τη δήλωση για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Ε, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Πέρασε η δήλωση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία και θέλω να ευχαριστήσω Τίσω τους συντάκτες καθώς και τον Charles Στάνερ που βοήθησε να ενεργοποιήσουμε συναδέλφους στο Στρασβούργο κάθε φορά. Επίσης ευχαριστώ το γραφείο μου το οποίο βοήθησε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα στα θεωρία έχουμε μία ομάδα νέων από την ΝΕΠΟΜΑΚ, την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήρθαν εδώ για την ανακοίνωση αυτής της δήλωση. Από αυτούς τους νέους εξαρτάται το μέλλον. Η υποστήριξη αυτής της δήλωσης ανοίγει το Συνάδελφε, εμείς χαιρετίζουμε την παρούσα αντιπροσωπεία και για να σεβαστούμε αντίστοιχα το χρόνο το λόγο έχουμε και ο κύριος Παπαστάμκος που ήταν και ο πρώτος υπογράφων της προηγούμενης δήλωσης που επίσης υποστηρίχθηκε πλειοψηφικά. Συνάδελφε Παπαστάμκο. Των συναδέλφων κύριο Ζεύκα, Σούστα, Μίτσελ και Μπεναμίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που προσυπέγραψαν τη δήλωση ε, παριθμών 7. Θέλω να ελπίζω ότι το χειρό μήνυμα του κοινοβουλίου θα οθήσει την κομισιόν ώστε να ασκήσει περισσότερο αποτελεσματικά τη συντονιστική της αρμοδιότητα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, ψηφοφορίες. Έξι προτάσεων ψηφίσματος για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Κοινό ψήφισμα. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ψηφίζουμε συνολικά την πρόταση υπέρ, κατά,